να ζητήσω το, από το Κοινοβούλιο να καλέσει για τον τερματισμό του στίγματος του HIV. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ούτε αυτό ήταν διαδικαστικό, αλλά την απόλυτα δικαιολογημένο. Απόλυτα δικαιολογημένο. Περνάμε τώρα στην έκθεση Γκραπίνη. Ενωσιακός Τελωνιακό Κώδικα. Η κυρία Γραπίνη ζητήσε το λόγο. Συγγήτρια, παρακαλώ. Έχετε το λόγο, κυρία Γραπίνη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω